Κυρίες και κύριοι, να σας καλωσορίσω και πάλι. Βλέπω ότι πέφτει ο αριθμός των παρευρισκόντων και των ε, ακροατών μας. 27, πολιτική ανταγωνισμού 2008. Ε, ο κύριος Πιτικόφερ είναι ε, ε, εισηγητής και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι βέβαιος ότι όσοι δεν συμμετέχουν ε, ε, με την παρουσία τους εδώ στη συζήτηση αυτή, σίγουρα το κάνουν με το πνεύμα τους. Ε, όσον αφορά την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Σοφία Ινετφέλτ, που είναι η συγγήτρια από την πολιτική ομάδα Άλτε των φιλελευθέρων. Και εγώ υποβάλλω πρόταση γνωμοδότησης, η οποία περιέχει 7 σημεία που θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφερθούν σε μια τέτοια γνωμοδότηση. Καταρχήν, πιστεύω ότι θα πρέπει να επικροτήσουμε την έκθεση αυτή, ιδιαίτερα το τελικό κεφάλαιο για τους ε, καταναλωτές και τα καρτέλ και είναι προφανές ότι τα καρτέλ ε, είναι εις βάρος των καταναλωτών και γι' αυτό ήθελα να το τονίσω αυτό. Δεύτερον, να πω ότι όταν έγραφα την έκθεση αυτή υπέθετα ότι ε, το COP15 θα είχε τελείως άλλα αποτελέσματα από αυτά που είχε τελικά. Ε, επί της αρχής όμως νομίζω ότι είναι σωστό να θέσουμε το ερώτημα τι επιπτώσεις θα έχουν τέτοιες διεθνείς συμφωνίες στην ανταγωνιστικότητα και στον ανταγωνισμό. Τρίτον, θα ήθελα να προτείνω να συμπεριλάβουμε την έκκληση προς την Επιτροπή στην επόμενη έκθεσή της να αφιερώσει ειδικό κεφάλαιο στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό. Ένα τέτοιο ειδικό κεφάλαιο θεωρώ ότι είναι κατάλληλο μέσο να τονίσουμε ε, κάποιο θέμα και ιδιαίτερα τις δυσκολίες που υπάρχουν στον ανταγωνισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα τέτοιο ειδικό κεφάλαιο. Έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέταρτον, να εξετάσουμε το θέμα Εγώ γράφω με ποιο τρόπο τα διάφορα εθνικά συστήματα στήριξη του τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία δημιούργησαν στρέβλωση του ανταγωνισμού. σω ε, θα έπρεπε να το διατυπώσω πιο προσεκτικά. Αν και κατά πόσο. Ε, ίσως θα έπρεπε να λέω, ίσως είμαι υπερβολικά επικριτικός, αλλά ε, ε μας ενδιαφέρει η σχέση ανάμεσα στους παραγωγούς και στους ε, Ε, πολιτές και πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό. Ε, το πέμπτο σημείο έχει να κάνει με τον ενεργειακό τομέα. Στην Γερμανία ε, πραγματοποιείται συζήτηση αυτή τη στιγμή, πιθανότητα και σε άλλες χώρες, διότι η έλλειψη επενδύσεων στον τομέα των υποδομών μπορεί να παρακολύουν ή παρακολύουν τον ανταγωνισμό. Έκτον, ε, μιλάμε για τις δημόσιες συμβάσεις. Και αυτό το σημείο το τονίζουμε διότι υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων που οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Και επίσης ε, στο σημείο 6 λέμε ότι αυτό γίνεται επειδή τα κριτήρια για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνιστώσεις θα μπορούσαν να τολίσουν τον ανταγωνισμό προς την ε, καινοτομία. Και έβδομο, ε, για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών ε, πιστεύω ότι συνεχίζει παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής να υπάρχει έλλειψη ανταγωνισμού. Και έχουμε συμπεριλάβει σχετική διατύπωση. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις δραστηριότητες του νέου Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Μπέρεκ στους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, είπα ότι με ενδιαφέρει η συνεργασία. Ε, στο βαθμό που έλαβα παρατηρήσεις τις έχω συμπεριλάβει και ευχαρίστω θα ήθελα να σας καλέσω να συνεχίσουμε την συνεργασία. Έχω συζητήσει το σχέδιο του κειμένου αυτού με την κυρία Ινετφέλτ η οποία μου είπε ότι θα επικροτούσε μια τέτοια γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον συνάδελφο Μπίτι Κόφερ για τη γνωμοδότησή του. Είναι ιδιαίτερα εξαντλητικό το έγγραφο και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και για τη συνεργασία γιατί η πρότασή μου έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο έχω κάποια σχόλια. Πιστεύω θα πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον. Καταρχήν, για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια δεν ε, λειτουργεί ακόμη η νέα αγορά ενέργειας γιατί κάποιες χώρες όπως οι χώρες της ε, Βαλτικής είναι ε, απονομονωμένες από την υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό εφηδιασμό και σήμερα πληρώνουμε ακριβότερα την ενέργεια από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχουμε πλήρες υποδομές στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά αυτό για την ενέργεια. Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε την πρόταση της κατάλληλης χρηματοδότησης των ενεργειακών υποδομών, έτσι ώστε να μπορούν τα σχετικά προγράμματα να εφαρμοστούν εγκαίρο και η Κομισιόν να υποβάλει εκθέσεις για το τι συμβαίνει για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα που θέλει να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, υπάρχει υποστήριξη για καθαρές μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον. Υποστηρίζω την πρόταση του συντάκτη της γνωμοδότησης ότι η Κομισιόν θα πρέπει να διερευνήσει πώς ε, οι κανόνες ε, περί ε, δημοσίων συμβάσεων επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στα κράτη-μέλη. Εγώ νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εκπονήσει ομοιόμορφους κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι επικεντρώνεται ο ανταγωνισμός στην κυροτομία και ακολουθούνται κανόνες διαφανής. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλετε αυτό το λόγο από την Κομισιόν. Ο κύριος συγγνώμη, δεν σας είχα δει. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον αδελφό Μπουτικόφερ για τα θέματα που Δεν έχω πολλά να προσθέσω για κάθε σημείο. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το έκτο σημείο που λέει να ενσωματωθούν οι πρόσκλησεις για τη δήλωση ενδιαφέροντος και οι συνθήκε σε μια σειρά προτύπων και κριτηρίων που θα αναφέρονται στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό θα τροποποιήσει τον αναγνωσμό. Θέλει να το βάλει σε άλλο βάση και θα δώσει μια σημαντική ε, οντότητα. Και θα ήθελα να σας πω κάτι που ενοχλεί για τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, το ανταγωνισμό είναι ένα μέσο, δεν είναι αυτός ο σκοπός, μέσο συχνά χρήσιμο, αλλά μέσο πάντα. Και αν δω το παράδειγμα της χώρας μου της Γαλλίας, όπου υπερβολική βούληση για ανταγωνισμό παρεμπόδισε τη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε σε ποιο κόσμο ζούμε. Θα πρέπει να έχουμε πρωταθλητές βιομηχανικούς και υπηρεσιών στην Ευρώπη και γι' αυτό καμιά φορά δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο με Δηλαδή, εντάξει, να αρνηθούμε τα καρτέν, να τα καταπολεμήσουμε, αλλά από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου την ανάγκη ενδυνάμωσης του βιομηχανικού δυναμικού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και αυτό το κριτήριο να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή θέλει κάτι να πει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι πολύ πλήρης και πολύ χρήσιμη, διότι ασχολείται με τα θέματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την εκπόνηση της έκθεσης στο μέλλον. Σημειώνουμε το γεγονός ότι εκτιμάται το ότι έχουμε επικεντρωθεί σε ειδικά θέματα στην έκθεση και ότι ζητήσατε ε, στο μέλλον να συγκεντρωθούμε για παράδειγμα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η σχέση ανάμεσα στον ανταγωνισμό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκεται στον πυρήνα των εργασιών μας. Το βλέπετε αυτό, με... το βλέπετε αυτό στις πρωτοβουλίες ε, που έχουμε ε, συμπεριλάβει, όπως για παράδειγμα για τις κρατικές ενισχύσεις. Σημειώνουμε λοιπόν αυτά που θα ήθελε να δει το Κοινοβούλιο στην επόμενη έκθεση. Όσον αφορά τα άλλα στοιχεία που συζητήθηκαν, τα σημειώνουμε, είναι πολύ χρήσιμα και θα προσπαθήσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που ακούσαμε στην επόμενη μας έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. θέλει να απαντήσει. Ναι, πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρατηρήσω, έχοντας ακούσει αυτά που είχε να πει ο συνάδελφο Βέμπερ, δεν θα περίμενα να επικριθώ για ότι εξυμνώ τον ανταγωνισμό. Παρακαλώ να το πείτε ξεκάθαρα σε όλες τις χώρες και στη δική μου τη χώρα. Ότι μου φαίνεται περίεργο που επικρίνεται εδώ η Επιτροπή Γι' αυτό θα ήθελα να πω στον κύριο Βέβε ότι οπωσδήποτε συμφωνώ με τι προθέσει σα. Δεν πιστεύω που δεν είναι ότι θα πρέπει ούτε να θεωρήσουμε ότι είναι άγιος ο ανταγωνισμός, αλλά οι αγορές χρειαζόνται τάξη. Μια αγορά χωρίς δημοκρατική τάξη δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό πάντα έτσι ήταν. Και η ιδέα ότι οι αγορές από μόνες τους μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την τάξη δεν είναι μια ιδέα που με βρίσκει σύμφωνο. Και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε ποια είναι η τάξη που έχει κάθε αγορά. Και μέσα στα πλαίσια της ε, ε, τάξης αυτής να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και με, μέσω της πλήρους ενημέρωσης αυτής ε, θα υπάρχει εξασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, εγώ σας ευχαριστώ. Προθεσμία 2 Φεβρουαρίου και μόνο στα αγγλικά γιατί η διαδικασία είναι πάρα πολύ σύντομη. Δυστυχώ. Τι να κάνουμε. Επόμενο σημείο. Έκθεση για την πράσινη βίβλο της Επιτροπή για διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το θέμα αυτό, ο εμπειρογνώμονας μας είναι ο Giles Chichester. Er hat das Wort. thank you. Um, my colleague, Mrs. Gutierrez, Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφό μου, η κυρία Γκουτιέρε, η πρώην συνάδελφο. σε, από άλλη πολιτική ομάδα, μου ζήτησε να πάρει εκείνη τη θέση μου. Το υπο, ε, το, είμαι διατεθειμένος ε, αν υποσχεθεί να ε, κάνει γρήγορα τη δουλειά της, να αλλάξουμε τη σειρά δηλαδή. Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αν συμφωνείτε όλοι. Θα αλλάξουμε λοιπόν τη σειρά. Θα συζητήσουμε πρώτα την ε- Ευρωπαϊκή. Ο συνάδελφος Εντσιού έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ως συντάκτης της νομοδότησης ε, θα σας παρουσιάσω τώρα τα συμπεράσματά μου για να σας αναφέρω ποια είναι η ανάλυση μου και ποιες είναι οι προτάσεις μου για την Κομισιόν. Καταρχήν, να σας πω να μην λάβετε υπόψη τη διατύπωση της έκθεσης που έχει διανεμηθεί γιατί υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ των διάφορων, διαφοροποίησεις μεταξύ των διάφορων μεταφράσεων να σας πω ότι θα έπρεπε να βελτιωθεί ε, ο τρόπος λειτουργίας ε, της ιστοσελίδας, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή να μην ε, λειτουργεί ως πύλη, γιατί έτσι όπως λειτουργεί σήμερα ως πύλη, τελικά απλώς διευκολύνει την δημοσιότητα και τη διαφήμιση για ορισμένα έργα που βρίσκονται σε κάποιες άλλες βιβλιοθήκες, για τις οποίες όμως η πρόσβαση ε, πρέπει να γίνεται επιπληρωμή. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι και πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Δεν μπορούμε να δώσουμε διασφαλίσεις για τη μόνιμη διάθεση των έργων. Ούτε θεωρούμε και ότι μπορεί να είναι πάντοτε δωρεάν η πρόσβαση στα έργα που λέγονται out of print αν τα έργα αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα σε έναν ιδιωτικό σερβερ, ε, τότε μπορεί ο ιδιοκτήτης ε, του σερβερ αυτού να, ε, αυτής της να ζητήσει αμοιβή για την πρόσβαση. Επίσης, χρειαζόμαστε έναν οργανισμό ή μια επιτροπή υπό την ηγεσία της Κομισιόν και μια πρότυπη και σίγουρη μέθοδο ε, για να ε, διασφαλίζουμε το σεβασμό των δικαιωμάτων του δημιουργού για τα έργα που προστατεύονται από τέτοια δικαιώματα. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή καθώς περιλαμβάνει έργα ψηφιακής μορφής, είναι πολύ πιο μεγάλη ε, από ότι μία οποιαδήποτε βάση δεδομένων. Η πρόσβαση ε, σε πληροφορίες ποιοτικέ για τους πολίτες, αυτό διακυβεύεται εδώ. Και ένας τέτοιος οργανισμός μας επιτρέπει να έχουμε ε, καλύτερη γνώση των ευθυνών και κάτι τέτοιο μόνο μπορεί να συνεισφέρει στην ορθή λειτουργία. Θα πρέπει να οργανώσουμε το θέμα των πηγών των ψηφιακών πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί μόνο να διαχειριστεί την ενιαία, μπορεί να διασφαλίσει με την ενιαία διαχείριση του project. Επομένω, είναι απαραίτητο να γίνει μία μελέτη από την Κομισιόν για τι δυνατότητες δημιουργία, μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, αλλά και εθνικών υπηρεσιών ή οργανισμών που να διαχειρίζονται τη διαδικασία ψηφιοποίηση, Να διασφαλίσει το σεβασμό των δικαιωμάτων του δημιουργού και την αμοιβή των δημιουργών. Πρέπει ε, όλα τα κράτη-μέλη εκτός από τις ε, κάτω χώρες, μάλλον τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφα όλων των έργων που έχουν δημοσιευτεί. Αν ε, έχουμε ε, και ένα ψηφιακό αντίγραφο, τότε οι πληροφορίες μπορούν ε, να κυκλοφορούν πιο γρήγορα και πιο φτηνά. Θα πρέπει να προστίθεται το νέο υλικό και το νέο αυτό θα διατίθεται πιο γρήγορα στους πολίτες. Και η αποστολή των ψηφιακών ε, υλικών στην Ευρωπαϊκή θα πρέπει να γίνεται μόνο από τους κατόχους των δικαιωμάτων δημιουργού. θα πρέπει αυτό το υλικό να χρησιμοποιείται δωρεάν για τους φοιτητές, τους μαθητές και τους καθηγητές. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Αυτή η κοινωνική κατηγορία θα πρέπει να έχει προνόμια σε σχέση με την πρόσβαση στο υλικό αυτή της βάσης δεδομένων. Η ε, αρμόδια υπηρεσία που θα διορίσει η Κομισιόν θα πρέπει να διαχειρίζεται το project. Στη κατηγορία αυτή θα μπορούσαν ε, να δεθούν ε, ειδικοί λογαριασμοί στο διαδίκτυο μέσω των οποίων ε, θα μπορούσαν να δουν το υλικό αλλά δεν θα μπορούσαν να το σώσουν. Οι νέοι θα πρέπει να αφήσουμε μάλλον τους νέους προς τη γνώση γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαβάσουμε τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Και το πρόβλημα που αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι το εξής. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο μέσω του οποίου μπορούν οι βιβλιοθήκες ε, να ε, προβούν στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα πρέπει να απευθυνθούν σε άλλους οργανισμούς βάσει ορισμένων συμβάσεων συνεργασίας ε, για να διασφαλίσουν την απελευθέρωση του υλικού. Σήμερα δεν γνωρίζουμε πολλές φορές ποιος κατέχει τα δικαιώματα του δημιουργού και φυσικά αυτό έχει επίπτωση στην ίδια τη διαδικασία ε, γιατί ε, πολλές φορές έχουμε και πάρα πολλά παλιά έργα και υπάρχουν προβλήματα με τη διαχείριση. Το project Europeana βρίσκεται σήμερα στο στάδιο Β Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πολίτε σήμερα δεν το γνωρίζουν πολύ καλά. Όταν θα λειτουργεί πλήρω θα πρέπει να υπάρξουν δημοσιεύσει και εκστρατείες ενημέρωση ε, για το πρόγραμμα αυτό, γιατί μια υπηρεσία είναι καλή μόνο αν χρησιμοποιείται και αν ωφελεί του πολίτε. Αν οι πολίτε συνεχίζουν ε, να χρησιμοποιούν το Google Books γιατί είναι πιο απλό το σύστημα αυτό και είναι πιο γνωστό, τότε το δικό μα ε, project θα είναι άχρηστο και τελικά απλώς θα έχουμε απώλεια ευρωπαϊκών πόρων. Δεν ε, θα προσδώσει αξία ε, στην Ένωση παρά μόνο αν αποτελεί το πραγματικό πολιτιστικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και φυσικά είμαι έτοιμος να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κουτήρας Κορτίνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Στην προηγούμενη Ισπανική Προεδρία Συζητήσαμε το θέμα αυτό και μάλιστα στην Επιτροπή Πολιτισμού και είδαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να εργαστούμε ε, σε ένα θέμα πολιτισμού αν υπάρχει επικουρικότητα γιατί η Ευρώπη δυσκολεύεται να διαχειριστεί ένα θέμα ε, το οποίο ανήκει στην επικουρικότητα. Δηλαδή πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα προς καμία κατεύθυνση ευρωπαϊκά, Έτσι όπως ε, έχει σήμερα είναι ένα σχέδιο με καλές προθέσεις αλλά δεν έχει σχεδιαστεί σωστά εγώ άκουσα τι είπε ο κύριος εισηγητής, αλλά πρέπει να δούμε τα εξή. Καταρχήν, η ιδέα της Ευρωπαϊκή είναι να υπάρχει μια διαβούλευση βιβλίων στο διαδίκτυο και να ε, υπάρχει επαφή με όλες τις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. Δηλαδή, πρέπει να συνδυάσουμε πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα τέλειο και ποιοτικό συντονισμό και ταυτόχρονα ε, να διοχετεύουν οι χώρες τις πληροφορίες σε αυτό το δίκτυο Europeana. Εγώ ε, δεν ε, θα ήθελα να δημιουργηθούν υπηρεσίες τέτοιες σε κάθε χώρες γιατί νομίζω ότι θα υπάρχουν δυσκολίες συνεννόησης μεταξύ τους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον επικεφαλής οργανισμό και πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο όπου φτάνουν όλες οι πληροφορίες για να έχουμε καλύτερη ποιότητα και ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικού δικαίου αυτή η οντότητα. Δεν ε, ξέρω τι συμβαίνει στις κάτω χώρες. Ε, πολλές φορές ε, μεταμφιέζεται το ιδιωτικό με το δημόσιο. Έχουμε πρόβλημα όμως πολλές φορές με τις ερευνητικέ πληροφορίες. Τα πανεπιστήμια πληρώνουν έναν οργανισμό στην Ολλανδία για να διανέμει τα περιοδικά και στη συνέχεια οι ίδιοι οι συγγραφείς πρέπει να πληρώσουν για να αγοράσουν το άρθρο τους και να μπορούν να το διαβάσουν. Η Ευρωπαϊκή λύνει το πρόβλημα αυτό. Εδώ Ό,τι είναι δημόσιο πρέπει να είναι ανοιχτό, πρέπει να είναι καλής ποιότητας και πρέπει να έχουμε και μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ε, πολλές ε, χώρες θα πρέπει να συνεισφέρουν και μπορούμε σήμερα, ε, δεν μπορούμε σήμερα να ζητήσουμε από κανέναν ευθύνε γιατί δεν λειτουργεί καλά το project αυτό. Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα γιατί εγώ έχω εμπειρία καθώς ε, ήμουν αρμόδια για το συντονισμό του πολιτισμού σε μια ισπανική περιφέρεια. Να σας πω ότι λέμε ε, ότι κάθε δάσκαλος έχει το δικό του βιβλίο. Έτσι λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη ε, δυσκολία να αλλάξει το σύστημα καταλογοποίησης από τη μία χώρα στην άλλη. Εγώ θα έλεγα μέσω ενός συστήματος, έχουμε λόγω χάρη διάφορα συστήματα, το PDF και τα λοιπά, να μπορούμε να τοπλοποιήσουμε τα πράγματα. Η Ευρώπη, ε, στην Ευρώπη χρησιμοποιούμε το TIF και το JPG, αλλά ε, εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να ζητήσουμε να έχει κάθε χώρα μία γλώσσα διαδικτύου και να χρησιμοποιούν όλοι την ίδια γλώσσα. Έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία και από την άλλη νομίζω ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα νομικό σύστημα μπορούμε να δημιουργήσουμε όμως έναν επικεφαλής οργανισμό γιατί αν ε, αρχίζουμε εδώ να δημιουργούμε νομικά συστήματα τότε ε, ουσιαστικά θα βρούμε περισσότερες δυσκολίες. Yeah, να πω στο ρημάνο συνελεφό αυτοί που περισσότερο αντιστέκονται στον συντονισμό του πολιτισμού είναι οι παλιοί, η Γερμανία και η Γαλλία και αυτό είναι αλήθεια. Πολλές φορές ε, βρήκαμε τέτοια εμπόδια σε διάφορα project. Νομίζω λοιπόν ε, ότι εμείς πρέπει εδώ να είμαστε ικανοί να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε την επικουρικότητα. Και κοιτάξτε, λόγω της επικουρικότητας δεν μπορούμε ε, να αναχαιτήσουμε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο με εικόνες, βίντεο και βιβλίων και έργων που να είναι προσβάσιμο στους νέους. Ε, ήδη σήμερα έχουμε μια νεολαία αδαή η οποία περνάει όλο, όλη τη μέρα μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Ας, δώσουμε κάτι ενδιαφέρον στους νέους. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή και να απευθυνθώ και στον κύριο Τσίτσεστερ. Είστε κύριος γιατί είστε gentleman, γιατί πραγματικά να μου επιτρέψετε να έχω τόσο χρόνο να μιλήσω. Έτσι λοιπόν θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε τον επικεφαλής οργανισμό και θεωρώ ότι αυτός ο συντονισμός μπορεί να επιτευχθεί με πολύ λίγα χρήματα και ταυτόχρονα μπορούμε να έχουμε κοινή γλώσσα έτσι ώστε να έχουμε στην λιγότερη νομοθεσία και μεγαλύτερη συμβατότητα. Δηλαδή, ε, η Ευρωπαϊκή ε, να μην έχει λιγότερους αναγνώστες από άλλα. Είναι ένα πολύ μεγάλος ύφαλος ε, αυτός που πρέπει να ξεπεράσουμε. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βητικόφερ έχει το ζητήσει στο λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Έντσιου για την έκθεση αυτή που μας έβαλε. Θεωρώ ότι δύο θέματα είναι πολύ σημαντικά, όπως τα τονίζει και ο ίδιος. Το ένα είναι το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης και το δεύτερο, το τονίσατε ιδιαίτερα συνάδελφε, είναι, είναι η αγκαιότητα να κάνουμε διαφήμιση της Ευρωπαϊκής, να γίνει γνωστό και κατανοητό αυτό, γιατί πολλά μπορούμε να κάνουμε, αν δεν το κατανοήσει κανένας ότι το έχουμε κάνει, δεν θα ωφελήσει κανένα και αυτό πραγματικά πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω κάποια λίγα σημεία Μία δυσκολία του Ευρωπαϊκού μέχρι τώρα είναι ότι η συμμετοχή των κρατών μελών είναι πολύ διαφορετικά έντονη. Η Γαλλία ιδίω και η Γερμανία είναι που, εκείνες που συμβάλλουν σε μεγαλύτερο ποσοστό. Και σίγουρα θα ήταν σημαντικό, ακριβώς επειδή αυτό είναι ένα σχέδιο για την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης, να υπάρχει πιο ευρεία και ισορροπημένη συμμετοχή. Δεύτερον, υπάρχουν μια σειρά νομικών δυσκολιών. Παραδείγματο χάρη, όταν συμπεριληφθεί υλικό το οποίο ακόμα προστατεύεται από copyright, γιατί δεν θέλουμε να ανοίξουμε μια μαύρη τρύπα εδώ τον 20ο αιώνα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να επιληθεί. Όπως και το πρόβλημα και εκείνων των έργων που είναι αδύνατο ή πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν οι δικαιούχοι. Τρίτη παρατήρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, έχουμε μία χρηματοδότηση του σχεδίου αυτού που να εγγυηθεί την βιωσιμότητά του. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκθεσή σας σε ευχαριστώ. Εξ νόμιτος της Κομισιόν, ποιος θέλει το λόγο, ο κύριος Φόλμαν, η κυρία Ζέλη. Yeah, thank you, Chair. Um... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Europeana είναι αποτέλεσμα μιας συνεργασίας χωρίς προηγούμενο μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτιστικών ιδρυμάτων. Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, είναι μια ε, ε, δουλειά που ε, αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται, αποτελεί Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ε, πρωτότυπο, αλλά ήδη δίνει ε, πρόσβαση σε πάρα πολλά δεδομένα, όχι μόνο βιβλία, αλλά και χάρτες, οπτικοακουστικό υλικό και άλλα. Ο πολιτικός στόχος είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των ε, αντικειμένων στα οποία δίνει πρόσβαση στα 10 εκατομμύρια και μέσα στη, εντός του έτους ε, θα λανσαριστεί ένα, μια αναθεωρημένη εκδοχή της Europeana. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης, ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης και οι προτάσεις που έγιναν θίγουν μια σειρά από πολύ σημαντικά θέματα, όπως για παράδειγμα τη βελτιστοποίηση της ε, ψηφιοποίησης στα κράτη-μέλη, η χρήση ε, κοινών προτύπων ε, και η μακρόχρονη διατήρηση του υλικού. Τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ψηφιοποίηση και πολύ σημαντικό θέμα είναι το πώς μπορεί η Europeana να γίνει πιο γνωστή στο ευρύ κοινό. Η ίδια η ομάδα της Europeana είναι αρκετά προσεκτική αυτή τη στιγμή με τη δημοσιότητα, ε, δεδομένου ότι η, βιβλιοθήκη υπερίσκεται ακόμα σε στάδιο πιλωτικό. Υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις στην ε, γνωμοδότηση, αλλά θα ήθελα να πω και λίγα λόγια. Ε, η Ευρωπιάνα είναι οργανωμένη με αποκεντρωμένο τρόπο και τα διάφορα ιδρύματα διατηρούν την, ε, ε, ε, ευθύνη. Η να βοηθάει την πρόσβαση σε υλικό από άλλες χώρες. αλλά προτείνεται ένα πολύ πιο συγκεντρωμένο μοντέλο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Με νέο σχέδιο το οποίο είναι διαφορετικό από ό,τι έχει αποφασιστεί μέχρι τώρα συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου 2007 και μια σειρά ε, συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Επίσης αναφέρθηκε η ελεύθερη χρήση στον πολιτισμό. Ε, ήδη η Ευρωπαϊκή δίνει πρόσβαση σε ε, πολύ υλικό το οποίο δεν ε, καλύπτεται από ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Βέβαια, η πρόσβαση σε υλικό το οποίο προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο θα έπρεπε να είναι δυνατόν να υπάρχουν συμφωνίες ε, ε, ε, αδειοδότησης με τους κατόχους των δικαιωμάτων ή θα μπορούσαν να υπάρχουν σύνδεσμοι από την Europeana στις σελίδες όπου οι χρήστες θα πρέπει να αγοράσουν το υλικό τελικά. Κάποιες παρατηρήσεις έγιναν για τους κανόνες για το copyright. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξέτασε αυτά και μάλιστα υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Οκτωβρίου που ασχολείται αναλυτικά με το θέμα αυτό. Η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση. Κεντρική σημασία για το όλο εγχείρημα της Europeana είναι αυτό και θα το εξετάσουμε ε, μαζί με τα ε, κράτη-μέλη και την ομάδα της Europeana. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχει εδώ ειδική διαδικασία, επιταχυμένη διαδικασία, διότι Είχαμε δυσκολίες ε, στην ε, Επιτροπή Πολιτισμού. Γι' αυτό αποφασίσαμε από κοινού ε, η ψηφοφορία να γίνει 5 Οκτωβρίου και οι τροπολογίες να υποβληθούν αποκλειστικά στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε την επόμενη εβδομάδα. φτάνουμε τώρα στο σημείο 30. Έκθεση σχετικά με την πράσινη βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τώρα τον Giles Chichester για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νόμιζα ότι παραλίγο να την κλειτώσω. Βιολογικά απόβλητα. Πράσινη βίβλος της Επιτροπής. Είναι αρκετά παλιά, είναι από το 2008 και ε, ορίζονται τα απόβλητα ως ε, ε, βιοδιασπόμενα βιοδιασπόμενα ε, ε, απόβλητα από εστιατόρια, από ε, καταστάσεις κήπους κλπ. καθώς και άλλα βιολογικά απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αναφέρει και τι δεν συμπεριλαμβάνεται στα βιολογικά απόβλητα, όπως για παράδειγμα υπολείμματα από δάση. Μας λένε ότι τα βιολογικά απόβλητα στην Ευρώπη είναι ανάμεσα στα 76,5 εκατομμύρια τόνους και 102 εκατομμύρια τόνους. Ε, από δύο βασικές πηγές προέρχονται από πάρκα και κήπους από τη μία μεριά και από την άλλη απόβλητα κουζίνας από την άλλη. Υπάρχουν διαφορετικές ε, εθνικές πολιτικές οι οποίες ε, εφαρμόζονται στην διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων. Αναφέρονται κάποιες από τις ε, παρούσες ε, μεθόδους διαχείρισης όπως είναι η ξεχωριστή συλλογή, ένα σύστημα το οποίο γνωρίζω όλο και καλύτερα ε, στο σπίτι μας όπου πρέπει να χωρίσουμε τα σκουπίδια μας σε διάφορα δοχεία. Τρελαίνεται κανείς προσπαθώντας να βάλει τα σωστά σκουπίδια στο σωστό κουτάκι στο σωστοδοχείο. Έχουμε κατόπιν ε, τους ε, χώρους υγειονομικής ταφής. Ε, συμφωνούμε ότι αυτό είναι κάτι κακό. Έχουμε την καύση. Μερικοί από εμά θεωρούμε ότι είναι κάτι καλό. Αρκεί να... Δεδομένου... Αρκεί να χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Έχουμε βιολογική βιολογική διαχείριση, ε, μεταξύ άλλων την ε, κομποστοποίηση και αυτό είναι κάτι που γνωρίζω. Ε, στην εξοχή βάζουμε όλα τα σκουπίδια μας σε ένα δοχείο και αφήνουμε να σαπίσουν για να χρησιμοποιηθούν κατόπιν για να λιπάνουμε το χώμα. Είναι πολύ οικολογικός ο τρόπος αυτός. Μιλάμε για αναερόβια ε, ε, διαχείριση, τα βάζουμε όλα αυτά ε, σε ένα δοχείο, βάζουμε κάποιο ακίνδυνο χημικό και παράγεται έτσι ένα αέριο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί ενέργεια. Είναι και αυτός ένας τρόπος κομποστοποίησης. Επανέρχομαι λοιπόν στο σημείο που έχει να κάνει με τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στην διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Ε, τρεις κατηγορίες, τρεις ε, προσεγγίσεις ε, εντοπίστηκαν. Η καύση, κάποια κράτη-μέλη μεταφέρουν κάποια από τα απόβλητα από τους χώρους υγειονομικής ταφής στις εγκαταστάσεις καύσης. Έχουμε κατόπιν ανακύκλωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπω δεν αναφέρεται στην κατηγορία αυτή και έχουμε και τις χώρες που βασίζονται κυρίως στις χωματερές. Κανένα κράτος μέλος δεν αναφέρεται εκεί, ωστόσο νομίζω ότι πολλά ε, κράτη-μέλη ε, χρησιμοποιούν χωματερές. Δεν είμαστε υπέρ των χωματερών, θα πρέπει να βρούμε νέο τρόπο διαχείρισης των ε, αποβλήτων αυτών. η βασική πτυχή του θέματος αυτού για την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά βέβαια είναι πάντα ωραίο να μοιραζόμαστε τις θέσει μας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το εμάς ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτό το θέμα στη δική μας νομοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντο έχει εκπονήσει έκθεση στην οποία λέει ότι οι δυνατότητε παραγωγή ενέργειας ε, από ε, τα στερεά απόβλητα είναι 20 εκατομμύρια τόνοι αντίστοιχων ε, σε πετρελαίου το οποίο μέχρι το 2020 μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό λοιπόν αξίζει τον κόπο να το ενθαρρύνουμε, διότι έτσι ουσιαστικά με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Διότι μπορούμε να παραγούμε από τα απόβλητα και να παράγουμε ενέργεια. Έχει λοιπόν εκδώσει η ε, Επιτροπή την πράσινη αυτή βίβλο που περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις τις οποίες ε, ε, καλείται ο κόσμος να απαντήσει. Μόνο μία από αυτές θα πρέπει, ε, κατά τη γνώμη μου, να απαντηθεί, που έχει να κάνει με την ε, παραγωγή ενέργειας από απόβλητα και πιστεύω ότι η δική μας ομοδότηση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό το θέμα. Να στραφώ τώρα στους συναδέρφους μου και να τους καλέσω να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, να συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτή. Έχω αρχίσει τη συγγραφή μια, ε, σχεδίου γνωμοδότησης, ε, αλλά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχω δει υπάρχει ακόμα χρόνος να ενσωματώσω άλλες προτάσεις και θα είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς τους συναδέλφους εάν έχουν να υποβάλουν σχετικές προτάσεις εφόσον ε, αφορούν ε, κόσμιους τρόπους να χειριζόμαστε τα απόβλητα. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφος όλοι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι φιλική και κόσμια, γιατί δεν θέλω να με κυνηγάτε μετά με τα απόφλητα. Σας ευχαριστώ. Ε, αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σας. Πράγματι, η ενέργεια από τα απόβλητα είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, μας απασχολήσει. σημειώνω ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο έγγραφο της Κομισιόν, στο ε, δυναμικό της αναερο, ε, επεξεργασίας και που θα μας δώσει ένα ανεξάρτητο, ε, μια ανεξάρτητη πηγή καυσίμων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για οχήματα ή θα μπορέσουν να περάσουν ε, στην, ε, στους αγωγούς φυσικού αερίου και να χρησιμοποιηθούν εκεί. Υπάρχει όμως μία σειρά τεχνολογιών που αυτή τη στιγμή εξελίσσονται και μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πολύ καλύτερα τα απόβλητα για λόγους ενεργείας. Το είχαμε εξετάσει αυτό όταν εξετάσαμε την οδηγία για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Θα θυμόσαστε τότε ότι δώσαμε κάποια ειδικά σημεία για το θέμα αυτών των βιοκαυσίμων από απόβλητα. Και το βλέπω στην εκλογική μου περιφέρεια η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μία διαδικασία που δεν οδηγεί σε βιολογικό αέριο, αλλά στην παραγωγή εθανόλης, δευτέρας γενιάς εθανόλης δηλαδή, ανησυχώ ότι εάν δεν το λάβουμε υπόψη σε συζήτηση αυτή τη στιγμή, θα φτάσουμε σε, μία, σε έναν ορισμό τη ανώδυνση επεξεργασία των αποβλήτων, που θα αναφέρεται μόνο στην παραγωγή αερίου και δεν θα αναφέρεται σε άλλες δυνατότητες που υπάρχουν ή που ενδεχομένως θα υπάρχουν μετά αύριο. Θα πρέπει και αυτό να το λάβετε υπόψη σας ίσως, αν είναι δυνατόν. Θα σας ήμουν πολύ ευγνώμη αν μπορούσατε να το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μάνα Γιώνα σας ευχαριστώ πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την σαφή εικόνα που μας παρουσίασε για το θέμα αυτό. Συμφωνώ ότι οι περισσότερες ε, πτυχές αφορούν την ε, ε, Επιτροπή ΕΝΒ. Η δική μας όμως δικαιοδοσία αφορά το εξής. Διαβλέπω ότι οι ενδεχόμενες επιλογές για νέες ευκαιρίες επιχειρήσεων είναι πραγματικά της δικής μας δικαιοδοσίας. Όχι μόνο όσον αφορά τη χρήση ενέργειας, αλλά και τη χρήση πρώτων υλών και περιττέρω εξεργασία. Επίσης θα να αναφέρω και το εξής. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, όχι μόνο για τη χώρα μου τη Σλοβενία, αλλά και γενικά ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ότι οι πολίτες δεν θέλουν να έχουν εγκαταστάσεις κοντά τους που, εξετάζουν, που επεξεργάζονται συγγνώμη, τα απόβλητα. Θα πρέπει να κάνουμε τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα δείχνοντάς τους συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες εικόνες ότι εμείς δεν πρέπει να συγκεντρώσουμε τους χιλιάδες μόνο σε ενός τύπου εγκαταστάσεις αλλά διαφόρων ειδών, ότι δεν υπάρχει μία μόνο δυνατότητα, πολλές δυνατότητες και να τους πούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και η δική μας επιτροπή είναι εκείνη που θα το πει αυτό ξεκάθαρα. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα ήταν καλό να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι χρειάζονται αηφόρα κριτήρια για τη βιομάζα. Και βάσει των κριτηρίων αυτών θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το πώς θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας τα βιολογικά απόβλητα. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο όσον αφορά τις νέες ε, πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Από όσο καταλαβαίνω, ο στόχος της ε, πράσινης βίβλου αυτή είναι να εξετάσει κατά πόσον χρειάζονται κοινοτικά μέτρα. Από όσο καταλαβαίνω, η απόφαση του ποια θα είναι τελικά η τεχνολογία που, που θα ε, χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά, τα τοπικά εκάστοτε. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί τι θα επιβάλλουμε εκ των άνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο συνάδελφος. Köszönöm, elnök, Köszönöm, úr. Szeretnék hozzászólni Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ είμαι χημικός μηχανικός. Έχω ασχοληθεί με βιοτεχνολογία 30 χρόνια. Κάτι λοιπόν καταλαβαίνω από το θέμα αυτό, όπως μας είπε και ο κύριος Σίτσεστερ στην έκθεσή του. Εξετάζουμε εδώ το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Και απόβλητα από τα οποία θα έπρεπε να παράγουμε μόνο βιολογικό αέριο. Κατά βάση. δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ούτε λόγω της ε, τεχνολογίας που υπάρχει, ούτε λόγω του, ε, του υλικού. Θα πρέπει εκεί λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Βιοεθανόλη δεν είναι σωστό, θα πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με το βιοαέριο και το βιομεθάνιο. γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ μπορεί το στεγνό υλικό να ξαναχρησιμοποιηθεί και το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από ένα καθαρισμό. Δεν θερμαίνει τόσο καλά όσο το φυσικό αέριο εκτός αυτού χρησιμοποιείται πολύ τοπικά σε μία μικρή κομμόπολη, σε ένα τμήμα μιας πόλης. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό πάνω σε αυτό το θέμα. Θα συνεργαστώ ευχαρίστως με τον κύριο Τσίστας. Η Τέχνης Καβέρσκε, παραδείγματος χάρη, είναι μια εταιρεία στη Σουηδία που ασχολείται με τις διάφορες αυτές μεθόδους και θα ήταν καλό να, να μας απασχολήσει μόνο αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει η Κομισιά κάτι να πει? Όχι. Κύριε Τσίτσεστερ, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Ε, ναι, δύο λόγια, Πρόεδρε, με την άδειά σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συμβολή τους και να πω ότι πραγματικά προέβλεπα ότι θα αναφερόταν το θέμα του να μην αποκλειστούν κάποιες τεχνολογίες. Γιατί μου φαίνεται ότι πραγματικά είναι σημαντικό να αφήσουμε όλες τις δυνατότητες ανοιχτές. Και θα ήταν καλό έτσι να μπορούμε να εισάγουμε και ένα στοιχείο ανταγωνισμού. Είχα κατά νου λοιπόν να προσθέσω κάποια παράγραφο να λέει ότι τονίζει σημασία να μείνουμε ανοιχτέ όλε οι τεχνολογικέ δυνατότητε για την διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και η δημιουργία θέσεων αποσχόληση σε αυτόν τον τομέα. Ελπίζω αυτό να καλύπτει τις ανησυχίε τη κυρία Χολ και τη κυρία Γιόρνταν. Και επίσης συμφωνώ με την παρατήρηση της για τα ε, αηφόρα κριτήρια. Όμως, έχω την εντύπωση ότι στη βιομάζα, αλλά εδώ δεν μιλάμε για βιομάζα, αλλά βιολογικά απόβλητα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η βιομάζα παράγεται επί τούτου και μετά μετατρέπεται σε καύσιμο, ενέργεια, βιοθανόλ κλπ. Ενώ τα απόβλητα είναι απόβλητα, σκουπίδια δηλαδή. Και θα ακούσω με ενδιαφέρον ε, όσα έχετε να πείτε για τις άλλες τεχνολογίες και θα μπορέσω νομίζω να προετοιμάσω τώρα το σχέδιο έκθεσης για την επόμενη φορά και Ελπίζω έτσι να μην δημιουργήσουμε κι εμείς πολλά απόβλητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κι εγώ. Το επόμενο σημείο είναι η διασφάλιση προστασία των δικαιωμάτων εννοητή συνεργασία στην εσωτερική αγορά. Εισηγητή ο Παύλου Ριμπίχ. Ο συνάδελφο απουσιάζει, αλλά η συνάδελφο Γερασίλικ τον εκπροσωπεί και τη δίνει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρίμπιχ δεν είναι εδώ, δυστυχώς. Θα προσπαθήσω να τον αντικαταστήσω, αλλά βέβαια όχι 100%. Γιατί ε, δεν μπορώ εγώ να πω 100%, αντικατορίσω 100% τα σχολεία σου, απλώ θα πω την προετοιμασία για μένα. Βέβαια θα διαβάσω και τα δικά σα σχόλια. Θέλει να προτείνει στην Επιτροπή Νομικών Επιθέσεων να, περιλάβει τι ακόλουθες συστάσεις. Καταρχήν, να προθεθεί η διαθεσιμότητα των ε, ευρωπαϊκών αδειών για τα δικαιώματα διανοητικής διοκτησίας κατόπιν ως ε, ένα βήμα για την εσωτερική αγορά για τα δικαιώματα διανοητικής διοκτησίας ε, να επιτρέπεται να υπάρχει μια άδεια που να επιτρέπει το έργο να διανεμηθεί σε εκείνη την γλώσσα να προαχθεί η ουδετερότητα και τα δικαιώματα τα διανοητική διοκτησία να διανέμονται ανεξάρτητα από το φορμάτι ή την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και να υπάρχει δυνατότητα μετατροπή μεταξύ των διάφορων φορμάτων να υπάρχει ε, ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία, ε, καθώ ε, θα υπάρχει και διαφάνεια σε ό,τι αφορά του κατόχου των δικαιωμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξουν ε, αποτελεσματικές κυρώσεις όταν υπάρχει παραβίαση του copyright ε, και παραδείγματος χάρη να υπάρχουν Συνάδελφοι, οι διερμήσεις παρακολούν να διαβάσετε κάπως πιο αργά, γιατί δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν αλλιώς. Okay, then I will start again. Θα τα ξαναπώ λοιπόν. Θα ξεκινήσω από το σημείο 5 να υπάρξουν αποτελεσματικές κυρώσεις ε, για την παραβίαση του copyright ε, και ε, να αποζημιώνονται οι κάτοχοι των δικαιωμάτων και να υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, Μάλλον ένα προβλέπεται από τις υπηρεσίες ε, αποζημίωση δεν υπάρχουν παραβιάσεις δικαιωματικής διεκτησίας να, υπάρχουν, ε, να, να, ισχύει το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο ανταγωνισμού όπου χρειάζεται να υπάρξει μια αξιολόγηση του αντικτύπου σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής διεκτησίας ιδίως σε ό,τι αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτό σε κάθε μελέτη αντικτύπου. Και τελευταίο σημείο, να ε, το παρατηρητήριο παρακολούθησης ε, της παραχάρηξης ε, να εκπονήσει κριτήρια προκειμένου να παράξει συγκρίσιμα δεδομένα για την καταπολέμηση της πειρατείας και της παραχάραξης σε όλους τους τομείς. Θα ήθελα να δεν βλέπω κανένα συνάδελφο να, είναι, να ζητά το λόγο και οι σκιώτες συζητητές λείπουν όλοι. Αυτό βέβαια μας συντομεύει τη διαδικασία. Και η Κομισιόν ίσως δεν θέλει να πει τίποτα. Πολύ ωραία, θαυμάσια. Οπότε κλείνουμε το σημείο αυτό της μέσης διάταξης. Και θα ήθελα να περάσω τώρα στο σημείο 31 που έχουμε το ίδιο, ο εισηγητής δεν είναι εδώ. Και γι' αυτό και αυτό δεν θα το εξετάσουμε. Πάμε στα διάφορα. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα. Η επόμενη συνεδρίαση 4 Φεβρουαρίου. Το ξέρετε όμω ήδη. Και γι' αυτό σα ευχαριστώ. Λυπούμε πάρα πολύ που πρέπει να κλείσω τώρα τη συνεδρίαση και να σα αφήσω ελεύθερου. Σα ευχαριστώ. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, ο κύριο συνάδελφο ο έχει κάτι πολύ σημαντικό να πει. Δεν μπορούμε να κλείσουμε ακόμα τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να αφήσω να περάσει αυτή τη στιγμή χωρίς να σας συγχαρώ για το ότι ολοκληρώσετε τη μέσια διάταξη ε, μέσα ε, στο χρονικό διάστημα που είχαμε και μάλιστα νωρίτερα γιατί αναγνωρίζετε πόσο πιέζονται τα μέλη ε, από χρονικούς περιορισμούς. Έτσι λοιπόν ε, σας πούμε τα καλύτερα και σας τα αναγνωρίζω.